ιατρικό προσωπικό και ασθενοφόρα, εκατοντάδες σχολεία κλειστά και κατεστραμμένα. Μισθοφόροι στέλνονται καθημερινά εκεί. Δεν πρόκειται πλέον για πόλεμο χωρίς μαχητές, όπως το ονομάζαμε στην αρχή. Είναι πια ε, πόλεμος με μαχητές που μάλιστα προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες. Και αυτό που βλέπουμε είναι μια κλιμάκωση όπου οδηγεί σε αύξηση της τρομοκρατίας, ε, μεταναστεύσεις και περιφερειακή σταθιά. Ο ειδικό εκπρόσωπος του ΟΗΕ, ο κύριος Σαλαμέ, ήρθε στο Συμβούλιο την Παρασκευή και είπε ότι ποτέ σε καμία άλλη σύγκρουση στον κόσμο, στο παρελθόν, δεν έχουμε δει τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις. Από τον Απρίλιο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει συναντηθεί, έχει συνεδριάσει 15 φορές με θέμα τη Λιβύη και τις 15 φορές απέτυχε να ζητήσει ανακοχή. Μιλώ για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΑΕΕ. 15 φορές. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια ελπίδα ε, να τεθεί σε ισχύ η ανακοχή, η κατάπαυση του πυρός μάλλον. Ελπίζαμε χτες πολύ. Σήμερα το πρωί όμως μάθαμε ότι δεν επήλθε συμφωνία στη Μόσχα και ο στρατηγό Χαφτάρ έφυγε από τη Μόσχα, εγκατέλειψε τη Μόσχα χωρίς να δώσει την συμφωνία του για την κατάπαυση του πυρός. Επανλημμένος έχουμε πει ότι εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με περισσότερη ενότητα. Η Γερμανία θα ανακοινώσει σύντομα, αν δεν το έκανε ήδη. Πάντως πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί, αν δεν έχει ήδη ανακοινωθεί από τη Γερμανία, ε, την, ε, το συνέδριο της διαδικασίας του Βερολίνου το Φλεβα... το... σε μερικές μέρες. Θα γίνει μια προσπάθεια να πανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πλευρέ με κατάπαυση του πυρό. Θα είναι μια καλή ευκαιρία. Ο ειδικό εκπρόσωπο ε, ήρθε την Παρασκευή. Ο Πρωθυπουργό κ. Σάραντ ε, τη αναγνωρισμένη κυβέρνηση ήταν στι Βρυξέλλε. Επίση, ε, συναντήθηκε με τον κύριο Σασόλη και με τον κύριο Μισελ. Δεν καταφέρουμε να συνενθούμε με την άλλη πλευρά του στρατηγού Χαφτάρ συζητήσαμε με συναδέλφους ε, από άλλες χώρες της περιοχής. Όλοι εκφράζουν τις ίδιες ανησυχίες. Η Λιβύη ε, ξεφεύγει από τον έλεγχο. Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα γίνει κατάβαση πυρός ότι, και ότι η διάσκεψη του Βερολίνου θα λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή. Στο τελευταίο, στην τελευταία συνάντηση του Συμβουλίου ε, είπα ότι στηρίζω την διάσκεψη του Βερολίνου. Προσπάθησα να, να ταξιδέψω στη Λιβύη. Δεν έγινε δυνατό για λόγους ασφαλείας. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι αρνήθηκα το ταξίδι μου για λόγους ασφάλειας. Δεν... <clears throat> Ήταν μάλλον μεγάλη ισχυρή η, η βούληση να μας δεχτούν. Χρειάστηκε να συναντηθούμε εδώ στη Βρυξέλλες με το Σάρατζ, αλλά όχι με το Χαφτάρ διαθέτω πλέον την εντολή μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να έρθω σε επαφή με όλα τα μέρη αν επιτευχθεί κατάβαυση του πυρός και αν γίνει, επέλθει συμφωνία ε, για, το πλαίσιο ειρήνευσης. Θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον έλεγχο του εμπάργου όπλων και για τον έλεγχο της ε, σχέσης κατάβασης του πυρός. Δεν ξέρω όμως ποιος θα το κάνει αυτό στην πραγματικότητα. Ε, ξοδεύουμε πολλά λεφτά στη Λιβύη. Παραπάνω από 630 εκατομμύρια σε βοήθεια συνεργασία στα τελευταία πέντε χρόνια. Ε, η Αφρικανική Ένωση κατάφερε να εκενώσει πάνω από 5.000 άτομα ε, που, είχαν, ε, που βρίσκονταν σε κατάσταση κινδύνου και έστειλαν πάνω από 50.000 άτομα ξανά στις αιστείες τους με δική μας βοήθεια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν 700.000 άτομα από την υποσαχάριο Αφρική στη Λιβύη. Δεν θέλουν όλοι αυτοί να έρθουν στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν δουλειές και ζουν εκεί και θα μείνουν στη Λιβύη. Όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες βέβαια. Αλλά αν η κατάσταση επιδεινωθεί και δουν ότι είναι κατόρθωτο να παραμείνουν στη Λιβύη, μπορεί να προσπαθήσουν να περάσουν στην Ευρώπη. Οπότε άλλη μια απειλή παράνομης μετανάστευσης μέσω της κεντρικής Μεσογείου ε, από τη Λιβύη, εκεί όπου οι Τούρκοι και οι Ρώσοι έχουν ηγετικό ρόλο Μέχρι πριν από λίγο, Ρουσία και Τουρκία ήταν ανύπαρκτες στην Κεντρική Μεσόγειο. Τώρα είναι επικεφαλής και ηγούνται των διαβουλεύσεων. Πριν από πέντε χρόνια ήμασταν δραστήρια, αλλά ήμασταν μόνοι. Τώρα εξακολουθούμε να δραστηριοποιούμεθα, λίγος πολύ. Σίγουρα περισσότερο τώρα από ό,τι πριν από έξι μήνες, αλλά de facto οι Ρώσοι και οι Τούρκοι έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να επηρεάσουν τα πράγματα γιατί έχουν στρατό επιτόπου. Όχι μέσω τακτικού στρατού, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι τα όπλα ρέουν και η ροή τους αυξάνεται. Η Λιβύη είναι σαν ένας καρκίνος, ένα καρκίνωμα το οποίο κάνει μετάσταση στο Σάχελ. Και αυτό έχει σχέση με το γεγονός ότι μεγάλες ποσότητες όπλων στη Λιβύη μολύνουν και τη γύρω περιοχή. Οι μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι στο Σουδάν μάλλον πολλοί από το Σουδάν, την ε, Συρία και την Μέση Ανατολή ε, φτάνουν στη Λιβύη για να πολεμήσουν. Αυτή είναι η κατάσταση στη Λιβύη. Ίσως να έχουμε καλύτερα νέα τι επόμενε 24 ώρε, ίσω όχι. Σω οι Γερμανοί συγκαλέσουν τη διάσκεψη, ίσως όχι. Σω καταφέρουμε την κατάβαση του πυρό, ίσως όχι. Δεν το γνωρίζω. Ελπίζω ότι θα ανοίξει ένα παράδειγμα ευκαιρία. Η, η Λιβύη είναι μια πλούσια χώρα, μια από τι πιο πλούσιε χώρε τη Αφρικανική Υπήρου. Παρόλα τα, παρόλη την πολιετή πολεμική σύγκρουση, εξακολουθεί να είναι πλούσια και θα μπορούσε εξαιτία του μικρού της πληθυσμού να ζήσει μια, ε, σε ευημερία. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται στον ένατο χρόνο μιας ε, πολιτικ καταστροφικής πολιτικής κρίσης. Κανείς δεν πίστευε ότι θα ήταν εύκολο η Λιβύη να βγει από 40 χρόνια μιας τρομακτικής ε, δικτατορίας και ξαφνικά σαν αποθαύμα να γίνει σταθερή δημοκρατία. Το ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο. Κανένας όμως δεν φανταζόταν μια τέτοια καταστροφή, ένα τέτοιο όλεθρο. Και παρόλα αυτά θα μπορούσε να, ακόμα και να χειροτερεύσει η κατάσταση. Και για τους Λίβιους και για εμάς. Αν δεν προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτή τη σύγκρουση και να βρούμε μια πολιτική λύση με τη στήριξη των κρατών μελών και του Ευρωκοινοβουλίου προφανώς θα προσπαθήσω να κάνω αυτό ακριβώς. Ελπίζοντας ότι αυτή η ενεργοποίησή μας θα μας καταστήσει τμήμα της λύσης προκειμένου να παραμείνει ενωμένη η Λιβύη και να βρούμε μια ειρηνική λύση. Ε, πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, αλλά αυτό το μάντρα Ε, το λέγαμε για πολλά χρόνια και για την Συριακή σύγκρουση και για τον Συριακό πόλεμο και τελικά η λύση ήταν στρατιωτική. Οπότε ίσως και εδώ να μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεδομένου ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε στρατιωτική λύση, μπορούμε να οχυρωθούμε πίσω από την εντύπωση ότι από τον ισχυρισμό ότι δεν, υπάρχει στρατιωτική λύση. Στην Συρία όμως, μέσω της δράσης της Ρωσίας και της ε, Τουρκίας, η λύση ήταν στρατιωτική. Μπορεί το ίδιο να συμβεί και στη Λιβύη. Και αυτό πρέπει να αποτελέσει ανησυχία και αγωνία για όλους μας. Διότι δεν θα είναι ευχάριστο στις ακτές της Λιβύης να δημιουργηθεί μια σειρά από ρωσικές και τουρκικές ε, βάσεις απέναντι από την Ιταλία που με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχουν τις μεταναστευτικές ροές πλέον και από τη Συρία και από τη Βόρεια Αφρική. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σοβαρά. Ελπίζω θα έχουμε καλά νέα τις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα λόγια σας. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, στις διάφορες πολιτικές ομάδες. Ο βασικός ομιλητής του ΕΛΚ είναι ο κύριος Ντέιβιτ Μακάλιστερ. Παρακαλώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. ακούσαμε από τον το εκπρόσωπο στη Λιβύη. Αυτή τη στιγμή εκτελήσεται ένα πολιτικό δράμα και στρατιωτικό στο κατόφλι μας και αυτό το δράμα ε, για πάρα πολύ καιρό δεν γνώρισε την προσοχή που πρέπει. Από τον Απρίλιο που επελάβνει ο στρατηγός ε, Χαφτά ε, έχουμε πάνω από χίλιους νεκρούς, πάρα πολλούς εκτοπισμένους, πολλοί εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια, τα δύο τρίτα είναι γυναικόπαιδα. Είναι πολύ μεγάλη εκτακτή ανάγκη αν την Κυριακή υπογραφή η εκεχηρία είναι ένα βήμα προόδου, όμω ο λαός της χώρας χρειάζεται βιώσιμη και μόνιμη ειρήνη. Το ακούσαμε. Η γερμανική κυβέρνηση, ιδιαίτερα η καγκελάριο, υποστηρίζει εδώ και καιρό δραστηριότητες για μια βιώσιμη λύση, και, ε, για να ξανάρθει βιώσιμη ειρήνη. Και αυτή η διάσκεψη που θα γίνει την Κυριακή στο Βερολίνο, κύριε είπατε, ε, θα συνεισφέρει ενεργά προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι το εξή και ω εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν συζητούμε για πρώτη φορά για τη σύραξη αυτή. Όλες οι χώρες που ενέχονται άμεσα ή έμεσα θα πρέπει να φροντίσουν αυτό ο εμφύλιο πόλεμος να τερματιστεί και να επανέλθει η ειρήνη στη Λιβύη. Στο μέλλον θα πρέπει να είναι μια κυρίαρχη και ειρηνική χώρα. Και μέχρι να γίνει αυτό δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για την ανοικοδόμηση. Από εκεί και πέρα θα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση, ιδιαίτερα για την Ένωση, να δώσει την υποστήριξή της. Ευχαριστώ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Το λόγο έχει η κυρία Κάτι Πύρη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα ε, το γεγονός ότι τόσο προκεχωρημένη ώρα. Είσαστε εδώ και δείχνετε ότι παίρνετε πάρα πολύ σοβαρά τις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και παρότι έχω προετοιμάσει ομιλία, σας υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά θα ακούσω την παρέμβασή σας και θα κάνω πολιτικές παρατηρήσεις αντί να διαβάσω την ομιλία μου. Σήμερα το πρωί ο κύριος Χαφτάρ έφυγε από τις διαπραγματεύσεις χωρίς να υπογράψει τη Συμφωνία Πάψης Πυρός, ε, ε, αυτό που ε, ξεκίνησε την Κυριακή. Βέβαια αυτό είναι ένα πλήγμα για τη Λιβύη, για τους ανθρώπους, για τη σταθερότητα στο Σαχέλ. Τους τελευταίους εννέα μήνες 208 ε, άμαχοι και εξίσου πολλοί ε, πολεμιστές ε, πέθαναν, έχασαν τη ζωή τους. Βλέπουμε υπάρχει όλο μεγαλύτερη παρέμβαση, όπως και η απόφαση της Τουρκίας να στείλει στρατεύματα. Έτσι λοιπόν στη Λιβύη βλέπουμε να υπάρχει πάλι ένας πόλεμος διαντιπροσώπων και ε, πρέπει να εμποδίσουμε την περαιτέρω κλιμάκωση. Κύριε είπατε εκπρόσωπε, εγώ χαίρομαι που ε, καταβάλλετε προσπάθειες την προηγούμενη εβδομάδα και σας καλώ να συνεχίσετε να κάνετε ό,τι μπορείτε για να διευκολύνετε την ε, επιβολή της πάψης πυρός ε, η συνδιάσκεψη που προβλέπεται για την Κυριακή είναι λίγο κρίσιμη και όπως και εσείς και εμείς όλοι ελπίζουμε ότι τελικά θα λάβει χώρα. Και τελευταία μου παρατήρηση, οι Λίβοι ε, έχουν ε, δικαιούνται να υπάρχει ελπίδα να ανοικοδομηθεί η χώρα τους. Νομίζω ότι γι' αυτό αγωνίζονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και επόμενος ομιλητής, ο κύριος Χαβιέ Νάρτ. Ευχαριστώ κύριε Μπορέλτ. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Αλλά αυτό που μας εκπλήσει είναι η ίδια μας η έκπληξη. Γιατί οποιοδήποτε είχε ακούσει επί τόπου ε, τους ε, ενεχόμενους θα ήξερε ότι η σημερινή τραγωδία δεν είναι σημερινή, είναι εννιάχρονη. Και τώρα μας εκπλήσει ε, αυτό που συμβαίνει στην Τρίπολη. Μα αυτό άρχισε από τις αντιφάσεις που είχαμε στη συμφωνία Φραγκενστάιν μεταξύ δύο αντιφατικών δυνάμεων ο Σαράς δεν εκπροσωπεί κανέναν. Ούτε τον ε, ε Χαφτάρ ακούσαμε, ούτε τους βουλευτές. Το μόνο που ακούσαμε εδώ είναι υποτιθέμενη νομιμότητα, ανύπαρκτη στη Λιβύη. Ακούσαμε τους εκπρόβους του Φαγέτ Αλ Σαράς θεωρώντας ότι μιλούν εξ ονόματος της Λιβύης. Η Λιβύη μιλάει σήμερα με τα όσα συμβαίνουν εκεί. Εγώ είμαι απολύτως κατά του πολέμου αλλά πολύ φοβάμαι κύριε Μπορέλο ότι από το κακό στο χειρότερο θα είναι τα νέα που θα ακούμε. Και η κατάπαυση του πυρός δεν θα βοηθήσει. Υπάρχει στρατιωτική ανισορροπία που δεν θα φύγει με ωραία λόγια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει. Αυτή τη στιγμή μας ευνηδιάζουν η Τουρκία και η Ρωσία. Αλλά είναι εκεί γιατί απουσιάζει μονίμως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είμαστε στη μεταφυσική νομιμότητα του Φαγέτα Αλσαρά και δεν αφογραζόμαστε την πραγματικότητα επιτόπου. Θα πρέπει να έχουμε επαφές αποτελεσματικέ, ουσιαστικέ και διακριτικέ και αν κάνει του κεφαλιού της η Γαλλία και η Ιταλία τελικά θα αποδείξουμε πόσο ανύπαρκτοι και, και ασήμαντοι είμαστε. Και ωραίες εκθέσεις γράφουμε και προτάσεις κάνουμε. Ο κύριος Σατουρί παρακαλώ έχει το λόγο. Ναι, λειτουργεί το μικρόφωνο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν πρόκειται για να συνεισφέρουμε στην ειρήνη στη Λιβύη, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιροτίζει, ευχαριστεί, λυπάται, διαβουλεύεται. Μιλάει, πολύ μιλάει, αλλά λίγο δρά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική και η παραμικρή προσπάθεια να ε, συνεννοηθούν και να συντονιστούν τα κράτη-μέλη. Κύριε Πορέλ, σας ζητάμε μήπως να είστε ο εγγυητής της Ευρωπαϊκής Διεθνούς Ανυπαρξίας. Όχι ακριβώς, γιατί όταν πρόκειται να εξωτερικεύουμε τη διαχείριση ε, των ε, συνόρων μας ε, με μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκεί συνεισφέρουμε χαροπά. Και είμαστε και εμείς όλοι μας υπεύθυνοι για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λιβύη. Και κύριε Μπορέλ, ποτέ δεν είναι αργά για να υπάρξουν οι αξίες της Ευρώπης. θα πρέπει να έχουμε διπλωματική δράση επιτόπου για την κατάπαυση του πυρός και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας ε, βοηθήσουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, να τους συνοδέψουμε. Ε, έχει ε, ακόμα χρόνο η υπόθεση αυτή για να σταματήσουμε στις κρατήσεις και στις απάνθρωπες συνθήκες. Κυρία Φρίσκο, από την Ταυτότητα και Δημοκρατία. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Μπορέλη. Ε, στην είσοδο αυτού του Κοινοβουλίου ε, έχει γραφεί ότι 500 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίοι ψήφισαν γιατί θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δραστηριοποιηθεί για την ασφάλεια της Ευρώπης, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011 και εκείνη συνέβαλε στο να αλλάξει το καθεστώς στη Λιβύη, αλλά τώρα έχουμε ένα αποτυχημένο κράτος. Και ποιος θα κρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση που συνέβαλε και αυτή στο να υπάρχει ο ανθρώπινος πόνος. Βλέπουμε το ρόλο που παίζουν η Τουρκία, η Ρωσία και ε, περιμένουν και η Κίνα και η Σαδική Αραβία. Αυτό είναι το λυπηρό αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια για την κοινή εξωτερική πολιτική αλλά καμία εξωτερική πολιτική. Ε, στην Μεσόγειο βλέπουμε και πάλι να ε, διεξάγονται μάχες γιατί η Ευρώπη είναι Μεσόγειος τελικά. Είναι κάτι που πρέπει να διερωτηθούμε. Ο κύριος Τζαμπάσκι έχει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε είπατε εκπρόσωποι, συνάδελφοι. Κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Διότι η συμφωνία μεταξύ Σάρατς και Ερντοάν περιλαμβάνει όχι μόνο την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στην Λιβύη, αλλά και την δράση εναντίον της Κύπρου και του Ισραήλ. Ο Σάρατς και ο Ερντοάν μεταφέρουν τα της Συρίας στο Λίβανο, στη Λιβύη, συγγνώμη. Ε, αυτοί που πολέμησαν στην Σύρια μετακινούνται τώρα στη Λιβύη. Και οι δύο αυτοί καθιστούν την Λιβύη ξανά υποταγή. Ευχαριστώ κυρία Ντεμιρέλ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι κυρίες και κύριοι. Η κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη και μια σοβαρή πολιτική λύση είναι απαραίτητη. Το 2011 το Άτομο βομβάρδισε τη Λιβύη και έριξε τον κυρίαρχο Καντάφη. Αποτέλεσμα, πλήρες χάος. Ε, βίαιος πόλεμο πόλεμος και πόλεμος δια αντιπροσώπων ουσιαστικά. Αυτός ο νατοικός πόλεμος τώρα ε, έχει πολλούς φορείς στη Λιβύη δεν είναι μόνο οι περιφερειακές δυνάμεις. Εκεί συμμετέχουν πλέον σχεδόν όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γεωπολιτική, ζώνε επιρροής και εξουσία. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ο πόλεμος όμως για το λαό εκεί σημαίνει δεινά και θάνατο. Και κύριε Μπορέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί συζητάει, μην τυχόν και έρθουν οι πρόσφυγες τα περισσότερα κράτη-μέλη συνεργάζονται όμως με την κυβέρνηση Σαράζ, ο οποίος ε, τα έχει κάνει πλακάκια με κάτι πολιτοφυλακέ που υποτίθεται ότι είναι και ακτοφυλακή τη Λιβύης για να μην έρχονται εδώ πρόσφυγες. Αυτά κάνει η Ένωση. Εξαγωγέ όπλων σε όλα τα μέρη τα εμπόλεμα θα πρέπει να σταματήσουν. Όλες οι, εξωτερικέ εξωτερικές δυνάμεις θα πρέπει να αποσυρθούν. Μόνο έτσι θα έχουμε βιώσιμη ειρήνη στη Λιβύη και όχι περαιτέρω κλιμάκωση με κούρσα πολέμου και εξοπλισμών. Και αυτό δεν βοηθάει κανέναν ούτε στη Λιβύη ούτε πουθενά άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό ο κύριος Νικολάου Αλαβάνος, παρακαλώ. Όχι μόνο απούσα δεν είναι όπως λένε μερικοί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ΝΑΤΟ έχουν βαρύτατες ευθύνες για την υπεριαλιστική επέμβαση, τον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη, για το διαμελισμό της συρίας. οι συνέπειες είναι καταστροφικές για τους λαούς ενώ και σήμερα ξανά οι ανταγωνισμοί ευρωπαϊκής ένωσης ή νατο με ρωσία και κίνα με την εμπλοκή χωρών όπως η τουρκία η αίγυπτος και άλλες για τον έλεγχο της ενέργειας έχουν διαμορφώσει εκρηκτική κατάσταση στη λιβύη και στην περιοχή. σε αυτό το επικίνδυνο για τους λαούς περιβάλλον η αστική τάξη της τουρκίας και με το απαράδεκτο τουρκο λιβικό σύμφωνο επιδιώκει να χαράξει αυθαίρετα τα θαλάσσια σύνορα στη μεσόγειο το αφήγημα των ισχυρών συμμάχων της ελλάδας και ο εφησυχασμός που καλλιεργεί η ελληνική κυβέρνηση έχει χρεοκοπήσει. οι ηνωμένε πολιτείε ευρωπαϊκή ένωση και νάτο θεωρούν την τουρκία στρατηγικό εταίρο με τη στάση τους οξύνουν την επιθετικότητά της. απάντηση είναι η ένταση της συντονισμένης λαϊκής πάλης για καμιά αλλαγή συνόρων ενάντια στις ξένες βάσεις ενάντια στις υπεριαλιστικές ενώσεις για να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά με τη δική του εξουσία με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα. Ο πρόεδρος Ταγιάννη από το ΕΛ και ένα λεπτό παρακαλώ. Όλοι περιμένουμε τη συνάντηση κορυφή του Βερολίνου και ελπίζουμε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Εγώ βέβαια δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Δυστυχώ όμω σε αυτή τη φάση η Ευρώπη ήταν ανύπαρκτη, ανύπαρκτε οι διάφορε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έδωσαν την απαραίτητη υποστήριξη στον ύπατο εκπρόσωπο. Έλειψαν οι πολιτικέ πρωτοβουλίε, τίποτα δεν έγινε. Ε, το αποτέλεσμα λοιπόν το βλέπετε. Τι βλέπουμε, βλέπουμε τη Ρωσία και την Τουρκία που έχουν γίνει σε τις κατάστασεις όχι μόνο στη Λιβύη αλλά σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Οι κίνδυνοι είναι όλο και μεγαλύτεροι. Ας μην ξεχνάμε την τρομοκρατία, την ε, μετανάστευση όσο δεν λύνεται το πρόβλημα στη Λιβύη και μετά υπάρχει και το μεγάλο θέμα της ενέργειας. Η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύη ε, ε, που τάραξε την Ευρώπη δεν πάει στη σωστή κατεύθυνση. Βλέπουμε να υπάρχει ένας νέος αγωγός, ο Ίστμετ που θα ενώσει το Ισραήλ με την Κύπρο, την και θα πάει μέχρι ε, την Ευρώπη για να έχουμε ενεργειακή αυτάρκεια. Η Ευρώπη πρέπει να λάβει μέρος και για να προστατεύσει την ενεργειακή της αυτάρκεια, την αυτάρκεια όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος ε, Κοτσολίνα. Αλλά ε, να σας πω ότι είναι πολύ αργά και έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους δεν θα δώσω το λόγο στο Κάτστιά, για να μην περιμένουν άσκοπα οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Κοτσολίνο. Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις που παρουσίασε ο ύπατος εκπρόσωπος. Ε, κάθε ώρα που περνάει και ακόμα και τα τελευταία λεπτά έχουμε κάποιες ειδήσει σχετικά με τη συμμετοχή στη συνάντηση του Βερολίνου την Κυριακή. Ανησυχούμε πάρα πολύ. Ε, μερικές φορές ε, αισθανόμαστε τον κίνδυνο του ότι είμαστε άχρηστοι και αναποτελεσματικοί. Η μόνη λοιπόν ευκαιρία που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίσουμε την κατάσταση είναι η πολιτική. Και δεν πρέπει να αρνούμεθα να χαράσουμε πολιτική. Πρέπει να είναι σαφή η στόχη μα. Να ενισχύσουμε τι διπλωματικέ προσπάθειε. Να διασφαλίσουμε το ότι δεν θα υπάρχουν ε, αντιπαλότητε. Θα έχουμε κατάπαυση του πυρό. Να λάβει χώρα η συνάντηση στο Βερολίνο. Να προσφερθεί βοήθεια σε όλου αυτού του Λίβιου, του τόσου πολλού Λίβιου, κυρίω τα παιδιά που και αυτά είναι θύματα του ε, πολέμου. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις πολιτικές προϋποθέσεις και τις θεσμικές για να ενισχύσουμε την πραγματική εθνική κυριαρχία της Λιβύης. Να υπάρχει ένας, ε, μια εκφοβιστική δύναμη. Νομίζω αυτό πρέπει να επιδιώξουμε. Μια δύναμη η οποία θα βοηθήσει το διάλογο και την ειρήνη γιατί ε, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνο με διπλωματικές προσπάθειες αν δεν έχουμε μια ευρωπαϊκή δύναμη και αφήνουμε το πεδίο ανοιχτό σε άλλες δυνάμεις, θεσμικές και πολιτικές. Εγώ νομίζω αυτό θα πρέπει να είναι το καθήκον μας αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ας μην ξεχνάμε ότι διδραματίζουμε καθοριστικό ρόλο για το μέλλον της Ευρώπης. Παίζουμε αποφασιστική παρτίδα στη Λιβύη για το μέλλον της Ευρώπης, ολόκληρης Ευρώπης και δεν μπορεί να είναι μια παρτίδα που θα την παίζουν μόνο λίγα κράτη, η Ιταλία ή η Γαλλία αν θέλετε. Αυτή λοιπόν τη δουλειά πρέπει να κάνουμε και να στηρίξουμε τον ύπατη εκπρόσωπο, τον κύριο Μπορέλ, για να αναπτύξει αυτή τη δουλειά του με επιτυχία. Σας λέω, είμαστε σε μια σημαντική παρτίδα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ολόκληρη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γκρόσελη από το Ρινιού. Ε, υπάρχουν κοιλίδες στη, στη συνείδηση κάποιων κρατών που ήταν υπέρ της επέμβασης εναντίον του Καντάφη. Όλα αυτά έχουν γίνει εφιάλτης πια. Και αυτός ο εφιάλτης οδηγεί ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων να προσπαθήσουν να περάσουν παράνομα τη Μεσόγειο και να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους. Η Τουρκία που εξακολουθεί να είναι επισήμω ε, υποψήφια χώρα έχει ξεκινήσει στρατιωτική εκστρατεία εκεί. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα δικά μα στρατηγικά συμφέροντα στη Μεσόγειο και τη Λιβύη. Η τουρκική παρέμβαση και η ρωσική παρέμβαση, αν ληφθούν υπόψη, μαζί με τα στρατιωτικά γυμνάσια στην Αίγυπτο, βλέπουμε προβλήματα που μπορούν να βγουν σύντομα από τα σύνορα της Λιβύης. Θα πρέπει να δράσουμε πολιτικά και οικονομικά αυστηρά και θα πρέπει οι δυνάμεις, οι εξωτερικές δυνάμεις να αποσυρθούν από τη Λιβύη, να ξεκινήσει μια πολιτική διαδικασία που θα φέρει ειρήνη και σταθερότητα στη χώρα και την περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μάρκ από τους ε, Πρεσένους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μπορέλ για όλα αυτά που μας είπατε και για τις προσπάθειές σας να επιτύχετε την ειρήνη στη Λιβύη. Νομίζω κανείς θεωρεί ότι είναι εύκολο να, έρθει, να επέλθει η ειρήνη ε, στη Λιβύη από το 2014 32.600 άνθρωποι πνίγηκαν στη Μεσόγειο και διερωτώμε με αν τελικά οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν τι θα μας πείραζε αυτό εγώ πήγα στη Μεσόγειο ε, σε επιχειρήσεις διάσωσης και αν μιλήσει κανείς επιτόπου με τους ανθρώπους ε, θα διαπιστώσει ότι στη Λιβύη οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι και είναι παντελώς απαράδεκτο απάνθρωπο το ότι εμείς ως Ευρώπη συμβάλλουμε στο ότι αυτοί οι άνθρωποι άνθρωποι κινδυνεύοντα τη ζωή του προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τι γίνεται, του ξαναπηγαίνουμε πίσω στον πόλεμο. Και διαρωτώ γιατί έπρεπε να στείλουμε στη Λιβύη περισσότερες περιπολίες, σκάφη περιπολίες από σκάφη διάσωσης. Ε, συζητάμε εδώ, αλλά δεν κάνουμε τίποτα έτσι ώστε να μπορούμε να σώσουμε τουλάχιστον του ανθρώπου εκείνου που φεύγουν από τον πόλεμο, από του ε, καταβλισμούς στη Λιβύη. Νομίζω θα μπορούσαμε να διασώσουμε περισσότερους ανθρώπους στη Μεσόγειο και τελικά αυτό είναι και το καθήκον που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τιερή Μαχιανή, για ένα λεπτό από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Οι δυτικέ δυνάμει παρενέβησαν στην Λιβύη και χειροτέρευσαν τα πράγματα. Οι γείτονε τη. Ε, ε, το ίδιο και οι γείτονε από τι χώρε Αφρική. Ε, τη στιγμή, αυτή τη στιγμή η χώρα είναι ξανά διχασμένη και πολλές ε, δυνάμεις ε, προσπαθούν να ε, πάρουν το πάνω χέρι και να ελέγξουν τις ροές από την Αφρική προς την Ευρώπη. Ο κ. Σαράτζ έκανε μια γύρο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τελευταία και οι τουρκικές δυνάμεις βρίσκονται στο πλευρό του αυτή τη στιγμή. Mm. Ο πρόεδρος Ερντοάν γίνεται de facto ο ισχυρός άνδρας και στην Συρία και στη Λιβύη και ελέγχει κατά κάποιο τρόπο τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Πώς μπορούμε να επιτρέψουμε στην αφέλειά μας να επικρατήσει. Η λύση θα είναι τελικά μάλλον στρατιωτική και εμείς θα είμαστε απόντες. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να είμαστε παρόντες σήμερα για να βοηθήσουμε τους Γάλλους στρατιώτες που βρίσκονται μόνοι τους και πολεμούν τον Ισλαμισμό στην υποσαχάρια περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κύριο ε, Φράγκος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμενος εδώ και εκπροσωπώντας την Ελλάδα, δεν μπορώ παρά να μην σταθώ στην ανάμειξη της Τουρκίας στην Λιβύη. Έχουμε καταλάβει που αποσκοπεί η ανάμειξη της Τουρκίας στην Λιβύη. Μήπως υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που πιστεύει όλες αυτές τις ανοησίε του Ερντογάν περί εφαρμογής του δικαίου. αν κοιτάξει κάποιος μόνο το πρόσφατο παρελθόν της τουρκίας μόνο εγκλήματα θα δει σφαγή χιλιάδων κούρδων στη συρία παράνομες γεωτρήσεις στην κύπρο καθημερινή παραβίαση των ελληνικών συνόρων και τώρα αποστέλει παράνομα μισθοφόρους τζιχαντιστές και όπλα στη λιβύη. είναι ξεκάθαρη η επιθυμία του ερντογάν να διεκδικήσει παράνομα ΑΟΣ μέσω της λιβύης σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών εθνικών δικαιωμάτων αυτό το γνωρίζει η ευρωπαϊκή ένωση. ως πότε η ευρωπαϊκή ένωση θα στηρίζει οικονομικά και πολιτικά τον εγκληματία ερντογάν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καστάλντο, κύριε Αντιπρόεδρε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε είπατε εκπρόσωπο, η χθεσινή συνάντηση στη Μόσχα με την, παράταση, με την παρουσία των Σαράσου και Χαπτάρ έδωσε δύο σαφή μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι ε, παρά τις ε, διπλωματικές πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τα διάφορα κράτη-μέλη, τελικά δεν προέκυψε καμία σαφή εξέλιξη. Προσπαθήσαμε να παίξουμε τον ρόλο που έπρεπε να παίξουμε, αλλά τι έγινε, μας πρόλαβαν η Ρωσία και η Τουρκία στην περίπτωση της Λιβύης έχουν βέβαια τα δικά τους συμφέροντα και αυτό που παίζει ρόλο είναι καταρχήν να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Σήμερα δυστυχώς ο Χαφτάρ επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπογράφει. Άρα δηλαδή αυτό ε, δίνει ίσως κάποια ευκαιρία να επέμβουμε. Αν θέλουμε να μην υπάρχει πάλι μια κατάσταση Συρίας θα πρέπει την Κυριακή να πάμε στο Βερολίνο να παρουσιάσουμε μια νέα πρόταση ε, μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως με το δικό μου, με τις χώρες της γειτονίας, την Ισία, Αλγερία. Ε, έχουμε τους εκπροσώπους του Ισλαμικού λαού, γιατί όλοι αυτοί υποφέρουν με αυτό τον πόλεμο ε, διαντιπροσώπων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε ε, πραγματικά να συμβάλλουμε στο να αφοπλίσουμε τις πολιτοφυλακές. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος το οποίο έλαβε χώρα το 2011. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε μπλε κάρτα. Τη δέχεστε. Παρακαλώ, κύριε Μαυρίδη. Σέβομαι πάρα Σα έχω γνωρίσει καλά και στην προηγούμενη πενταετία και ήθελα να μα πείτε την άποψή σα για το εξή θέμα για να το ακούσει και ο κύριο Μπορέλ. Το καθεστώ στην Τρίπολη τη Λιβύης έχει προβεί σε μια συμφωνία με τον ερντογάν με βάση την οποία η τουρκία απέκτησε λέει αως στην ανατολική μεσόγειο με ένα κράτος τόσο πολύ μακριά ώστε περίπου να μπορούσε η τουρκία να ρυθμίσει αως και με την κώστα ρίκα. τι θα συμβουλεύατε τον κύριο μπορέλ να πράξει για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική επιθετικότητα η οποία στις επόμενες εβδομάδες λέει ότι θα στείλει ερευνητικά πλοία εκεί στο μέρος που είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα της ελλάδας όπως έπραξε και στην κυπριακή ΑΟΣ. Αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, αγαπητέ Κώστα, όπως ε, ε, πολύ σωστά γνωρίζεις, εγώ έχω επικρίνει πολλές φορές αυτή τη συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας που δεν ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και κυρίως ε, θέτει σε κίνδυνο τα νόμιμα συμφέροντα κρατών μελών όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Δεν πιστεύω ότι αυτή η μονομερής στάση μπορεί να γίνει ανεκτή κυρίως λόγω του ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς βλέπουμε ότι κλιμακώνεται η ένταση στη Λιβύη. Ε, εκεί παίζονται γεωπολιτικά παιχνίδια. Ε, ως εκ τούτου θα πρέπει να αποφευθεί ε, πάση θυσία υπεραιτέρω κλιμάκωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι περισσότερο παρούσα. Θέλω να δείξω εμπιστοσύνη στον είπα το εκπρόσωπο ότι θα συζητηθούν την Κυριακή συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Να προλάβουμε καταστάσεις πριν είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Μεϊμαράκης από το ΕΛΚ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ προσοχή την ανάλυση που έκανε ο κύριος Μπορέλ και πρέπει να σας πω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ δεν είμαστε αναλυτές, είμαστε πολιτικοί και οι πολιτικοί πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις. Πρέπει να μην είμαστε θεατές και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις αλλά να παρεμβαίνουμε στις εξελίξεις και να δίνουμε λύσεις γιατί αυτό θέλουν οι πολίτες που αγωνιούν και ανησυχούν για την ειρήνη στην περιοχή. από την ανάλυση που μας έκανε φάνηκε ότι η ρωσία και η τουρκία είναι οι κυρίαρχες δυνάμεις στην περιοχή. γιατί είναι; γιατί εμείς αφήσαμε ένα κενό το οποίο ήρθαν και κάλυψαν. κατά συνέπεια πρέπει εδώ ο κύριος μπορέλ να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ε, ειρήνη στην περιοχή και εμείς όλοι θα στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. και το κύριο πρόβλημα είναι η τουρκία η συμπεριφορά της τουρκίας είναι αυτή που δημιουργεί και απαξιώνει τις αρχές και τις αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης και μας δείχνει με την προκλητικότητά της ότι θέλει να ακολουθήσει τη δικιά της πορεία. αμφισβητεί λοιπόν κανείς σήμερα ότι αυτή η συμπεριφορά είναι αυτή προκλητική που μας αναγκάζει κιόλα και μας ε, προτρέπει στο να επέμβουμε για να υπάρχει ειρήνη. εμείς θα στηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίες που θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση και η ευρώπη πρέπει να δείξει ότι υπάρχει και είναι παρούσα στην στην περιοχή για την ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σπίτσουλα για ένα λεπτό από τους σοσιαλιστές. Ένα ε, λεπτό και κάτι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το θέμα αυτό είναι κρισιμότατο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει επισκιαστεί δυστυχώς από άλλα θέματα όπως το Ιράκ και το Ιράν τελευταία. Ε, αυτή τη στιγμή η Τουρκία που επισήμως είναι σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ συντονίζεται με άλλες, περιοχές, με άλλες χώρες της γειτονιά μας και ενώ η Ρωσία παραβιάζει ε, κατά σύστημα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ε, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να μην βρίσκουν μια κοινή θέση σε ό,τι αφορά τη Λιβύη. Η στρατιωτική παρέμβαση ίσως ε, δεν θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα του χάου στην Λιβύη, μπορεί ενδεχομένω μάλιστα να το αυξήσει. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε στη μεταναστευτική πολιτική όμως εμείς, πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις χώρες της γειτονίας μας. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις ε, δράσεις των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ. Ζημριοκ από το ID. Πρόεδρε, στρατιωτικά ε, δυνάμεις στην ε, Λιβύη. Μετά τη συμφωνία ε, για τους πρόσφυγες είναι η επόμενη κίνηση στο σκάκι που παίζει ο Ερντοάν με την Ευρώπη για το μεταναστευτικό. είμαστε ρεαλιστές. Σήμερα δεν πρωταγωνιστούμε εμείς εκεί. Δεν έχουμε το πάνω χέρι την κρίση του μεταναστευτικού και δεν αποφασίζουμε εμείς, αλλά ο Ερντογάν για τις μεταναστευτικές οδούς και αποφασίζει πόσο μεγάλη θα είναι η μαζική μετανάστευση. Πολύ εύκολα μπορεί να μας απειλήσει με το επόμενο μεταναστευτικό ρεύμα και αρχίζουμε να φοβόμαστε. Και τώρα με τη Λιβύη θέλει να ελέγξει εκείνη την Αφρικανική χώρα από όπου έρχονται οι περισσότεροι ε, παράνομοι μετανάστες προς την Ευρώπη. Συμπέρασμα, ο Ερδογάν μας έχει στο χέρι και μπορεί να μας εκβιάζει ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την οικονομική και στρατιωτική μας ισχύ και να αποδειχθούμε ε, εισάξη. Ε, αντίπαλοι. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί για να τερματιστεί η παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη, ε, να καταγγελθεί η συμφωνία για τους πρόσφυγες και να πάρουμε στα χέρια μας την επιφύλαξη των συνόρων μας. Από το ECR, ο κύριος Φιντάντζα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο πόλεμος διαντιπροσώπων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Λιβύη αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ασυνέπεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, και αυτά που είπε ο κύριος Μπορέλ σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μνημείο ανικανότητας. Βλέπουμε ότι ορισμένες χώρες, στο παρελθόν η γαλλική κυβέρνηση από το 2011 έπαιξε στην ε, Τρίπολη ε, και έτσι προκάλεσαν την κρίση. Η Τουρκία έχει τις δικαδικά της σχέδια, τα νέα Οθωμανικά ε, και ενώ αυτά γίνονται στη γειτονιά μας βλέπουμε ότι η Ευρώπη είναι απούσα. Είναι απούσα, απόν και, το, και, απούσα και η Ιταλική κυβέρνηση, ε, ενώ βλέπουμε ότι άλλα κράτη ε, προσπαθούν να παρέμβουν σε μια περιοχή που εμείς ασκούσαμε επιρροή. Λείπουν ακόμα ε, λίγες ημέρες για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση και να αποφύγουμε μια καταστροφή. Ο κύριος Λαγός, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Μου προκαλεί πραγματικά κατάπληξη και θυμώ ταυτόχρονα αυτό που άκουσα πριν από λίγο από τον κύριο μπορέλ παραδέχτηκε επίσημα ότι κουμάντο στην περιοχή κάνει η ρωσία και η τουρκία και ειδικά όταν μιλάμε για την τουρκία μιλάμε για ένα κράτο δολοφόνο για ένα κράτο το οποίο είναι βαμμένο με το αίμα αθώων εκατομμυρίων αθώων πολιτών από πολλέ χώρε και εμεί αυτή τη στιγμή κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και λέμε επίση ότι είναι αναγνωρισμένη η κυβέρνηση του αλ σάρατ. Η κυβέρνηση αυτή που έρχεται σε σύμπραξη με τον ερντογάν με τον δολοφόνο ερντογάν που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ο ερντογάν έχει πάρει δυνάμει τζιχαντιστών από αυτού που πολεμούσαν στη συρία και τι έχει μεταφέρει στην λιβύη έχει μεταφέρει το πρόβλημα ακόμα πιο κοντά λοιπόν στην ευρώπη δίνει όπλα με παράνομο τρόπο στον σάρατ και εμεί αυτόν εδώ λέμε ότι τον αναγνωρίζουμε. αυτό είναι απαράδεκτο και επίση είναι ντροπιαστικό για την ελληνική κυβέρνηση να ανέχεται αυτή τη στιγμή στη συνδιάσκεψη που θα γίνει σε λίγε μέρε στο βερολίνο να είναι παρόν το κονγκό να είναι παρούσα η Αλγερία και να απουσιάζει η Ελλάδα. Όμω και εσεί είναι ντροπιαστικό αυτό που κάνετε στη χώρα μου. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να υπερασπίζεστε την Τουρκία και να αδικείτε την Ελλάδα. Και στο κάτω-κάτω η Ελλάδα είναι ένα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ είναι δυνατόν να αδικείτε συνεχώ υπέρ τη Τουρκία. Να ξέρετε κάτι, δεν είμαστε διαθετημένοι να παρατήσουμε την Ελλάδα και δεν είμαστε διατεθειμένοι να σταματήσουμε τον αγώνα. Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μα με οποιοδήποτε τίμημα. Και ό,τι ξέρατε μέχρι τώρα για κάποιου ανθρώπου που σκύβαν το κεφάλι, ξεχάσετε από εμάς. Ευχαριστώ. Κύριος Κάρας, αντιπρόεδρος, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Κύριε Αντιπρόεδρε, όλο και σαφέστερο γίνεται από τις απόψινές συζητήσεις, το απόγευμα και τώρα τόσο αργά, στις αιστείες ανάφλεξης και κρίσης σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουμε ρόλο, δεν παίζουμε ρόλο ακόμα και αν είναι στο κατόφλι μας. Και έχουμε την αίσθηση ότι ε, κάπως αμφιταλαντευόμαστε ανάμεσα στη δράση και την αδράνεια ε, στα λόγια και στα έργα. Εγώ δεν βλέπω πολιτική αποφασιστικότητα, πολιτικό όραμα και δράση και η Λιβύη είναι αντανάκλαση ε, της κατάστασης της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, μετανάστευσης, γειτονίας, εξωτερικής και πολιτικής ασφάλειας, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Και αυτό το κενό που ανέφερε ο κύριος Μεϊμαράκης έρχεται να το καλύψει η ε, Τουρκία με τη Ρωσία. Τώρα έχουμε μια ευκαιρία το Σαββατοκύριακο στη Σύνοδο Κορυφής του Βερολίνου να έχουμε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Παρακαλώ πείτε μας ότι θα έχουμε ένα ρόλο στο Βερολίνο να παίξουμε σημαίνοντα. Ευχαριστώ η Μαρία Ρενά από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Για ένα λεπτό. Η κατάσταση στη Λιβύη είναι απαράδεκτη και για τους αμάχους στη Λιβύη αλλά και επικίνδυνη για την περιφερειακή σταθερότητα, το Μαγκρέπ, το Σάχελ και βέβαια επικίνδυνη και για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αν προσθέσουμε και τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε. Ε, ακτιβιστές ε, δολοφονούνται ή εξαφανίζονται. Ο Σιαμ Σεργιουάκ που, ήταν, που είναι βουλευτή, έχει εξαφανιστεί πριν εδώ και έξι μήνες. Ε, άλλοι την χάνουν κακής μεταρρύθμισης. Ε, με τις ε, παρεμβάσεις της ε, Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Ρωσίας ε, όχι μόνο οι στρατιωτικοί παίρνουν την εξουσία αλλά περασπίζονται και ένα μοντέλο που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και η Ευρώπη έχει να παίξει ρόλο, ένα σημαντικό ρόλο σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο. Η διάσκεψη του Βερολίνου προφανώς, η διαμεσολάβηση μεταξύ όλων των παικτών και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας είναι ο ρόλος μας. Ευχαριστώ. Ε, και τώρα ε, επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Ασημακοπούλου από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παρακαλώ. Αδελφοί, είναι επιτακτική ανάγκη αλλά και υποχρέωση της Ευρώπης να διεκδικήσει έναν ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις στη Λιβύη. Γιατί πρώτοι εμείς θα υποστούμε εδώ στην Ευρώπη τις συνέπειες, οπότε καλωσορίζουμε την ειρηνευτική διαδικασία του Βερολίνου, την οποία η Τουρκία τορπιλίζει με την επιμονή της να εφαρμοστεί το άκυρο και ανυπόστατο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της τουρκίας και της κυβέρνησης της τρίπολης με αποτέλεσμα να έχει αποχωρήσει σήμερα ο χαφτάρ από το τραπέζι των συνομιλιών. η ευρωπαϊκή ένωση έχει πάρει ξεκάθαρη θέση ότι το μνημόνιο της τουρκίας με την κυβέρνηση της τρίπολης παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και δεν παράγει οποιοδήποτε ένομο αποτέλεσμα. πρέπει λοιπόν κύριε μπορέλ παρά αυτά να απαιτήσετε από τον ερντογάν και τον σάρας να σκίσουν το παράνομο μνημόνιο τουρκίας τρίπολης ως ελάχιστη ένδειξη προσήλωσης στην ειρήνη και στην ασφάλεια της ανατολικής μεσογείου. οι αναπάντητες τουρκικές προκλήσεις δεν απειλούν πλέον μόνο την ειρήνη αλλά πλήττουν την αξιοπιστία της ευρώπης και εν τέλει υποθάλπουν το ίδιο της το μέλλον. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ε, ε, ε, κυρία σε Σεσάρτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Κυρία Πρόεδρε, η διαχείριση της ελληνικής ε, κρίσης αποδεικνύει την ανεπάρκεια της Ιταλικής κυβέρνησης σε ένα τόσο λεπτό και στρατηγικό θέμα. Βεβαίω όλα ξεκίνησαν με την καθαίρεση του Γκαντάφη πριν από 10 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια η Ευρώπη επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε ένα κενό, χώθηκαν εκεί η Ρωσία και η Τουρκία και παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην σκακέρα της Μεσογείου. Η Άγκυρα παίρνει τα κλειδιά της εισόδου σε αυτή την περιοχή. Η Λιβύη, ε, η Ιταλία έχει συμφέροντα στη Λιβύη. Ε, τα γεγονότα όμως ε, είναι αμήλικτα. Η Ιταλική κυβέρνηση είναι ανίκανη στην εξωτερική πολιτική και αυτό πιστοποιήθηκε για άλλη μια φορά. Η κατάπαυση του πυρός δεν υπογράφηκε στη Μόσχα. Ίσως θα έπρεπε να υπογραφεί στη Ρώμη, ούτε και αυτό συνέβη. Και τώρα πλέον όλος ο κόσμος περιμένει την υπογραφή στο Βερολίνο. Αν η Ευρώπη για άλλη μια φορά αποτύχει, ε, θα είναι άλλο ένα βήμα προς τα, πίσω, προς τα πίσω σε μια διεθνή πολιτική που μας βλέπει ότι είμαστε όλο και πιο περιφερειακοί. Περιφερειακοί, με σχολεία. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Πισάπια. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, είπατε πολύ σωστά ότι στην Λιβύη τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και από τη σημερινή συζήτηση ε, προκύπτει ε, μια αντισόπιτη αλήθεια. Δυστυχώς ε, στη Λιβύη επικρατεί το μοντέλο Ερντογάν και το μοντέλο του Πούτιν. Έχουμε μεγάλες ευθύνε, φέρουμε ευθύνη, πρέπει να ξεπεράσουμε την ομοφωνία. Η ομοφωνία όμω αυτή πολλέ φορέ μα εμποδίζει να αντιδράσουμε αυτή, αυτές οι ίσες αποστάσεις ε, από τους δύο ε, στη Λιβύη μας εμποδίζει να προχωρήσουμε. Δεν θα υπάρξει ποτέ Λιβύη, ε, ειρήνη στη Λιβύη με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν καλές προθέσεις, αλλά καλές προθέσεις δεν πάβουν ένα πόλεμο. Πρέπει λοιπόν να επιβληθεί εμπάργο όπλων και θέλω να σας υπενθυμίσω τα λόγια του Τζον Κένεντι. Δεν θα πρέπει να έχουμε το φόβο του να διαπραγματευόμεθα, αλλά δεν πρέπει ποτέ να διαπραγματευόμεθα γιατί φοβόμαστε. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Λαντσίνη. Κύριε Πρόεδρε, στην Λιβύη, παρά τι δηλώσει προθέσεων, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην αποφασίσει και άφησε το πεδίο ελεύθερο στη, Ρωσία, στη Ρωσία και στην ε, Τουρκία. Ε, πρέπει, σα είπα και άλλε φορέ, ε, να απαγορευτούν ε, οι εξαγωγέ όπλων στην Τουρκία και σε άλλες χώρες. Δυστυχώς λοιπόν η κυβέρνηση της ε, Τρίπολης ε, διαπιστώνουμε ότι πλέον συνεργάζεται μόνο με τον Ερντογάν ε, για θέματα όπλων και σήμερα βλέπουμε ότι και ο Ερντογάν στέλνει τζιχαντιστές και κανονικά στρατεύματα στη Λιβύη. Αυτή η κατάσταση είναι επικίνδυνη, μπορεί να αποσταθροποιηθεί περαιτέρω η περιοχή, κυρίως να τεθούν σε κίνδυνο τα ιταλικά συμφέροντα. Μία τελευταία έρευνα του Associated Press σχετικά ε, για το πού κατευθύνονται τα χρήματα των Ευρωπαίων απέδειξε ότι ε, ένα μεγάλο τμήμα των χρημάτων που δόθηκαν για να σταθεροποιηθεί η περιοχή και να βελτιωθούν οι καταβλισμοί, τα χρήματα αυτά πάνε στη Λιβική ε, πολιτοφυλακή και στις εγκληματικές οργανώσεις. Αυτό δυστυχώς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιρροή της Ρωσίας και της Τουρκίας και αυτά όλα αποδεικνύουν το ότι αποτύχαμε στη Λιβύη. Ο κύριος Φουρλάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπορέλ, η κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Λιβύη δεν πρέπει να αφήνει κανένα αδιάφορο. Η Λιβύη σήμερα κινδυνεύει να μετατραπεί σε δεύτερη Συρία. Και αυτό γιατί κάποιε χώρε, όπω η Τουρκία, έχουν ηγεμονικέ τάσει στην περιοχή, κύριε Μπορέλ. Η Τουρκία έχει βάλει πόδι στη Λιβύη. Και εμεί παρακολουθούμε μη ξέροντα πώ να αντιδράσουμε, βαρώντα παλαμάκια. Ο φασίστα Ερτογάν κάνει ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή την ευρώπη. έχετε εντύπωση ότι θα πάτε στο βερολίνο θα πάρετε μια απόφαση την οποία θα σεβαστεί η τουρκία. Πεστε μου ποια απόφαση σεβάστηκε ή ποια συμφωνία η τουρκία και να συμφωνήσω μαζί σα. καθήκον μα είναι να παρακολουθούμε τι όποιε εξελίξει στην προσφυγική κρίση και την πιθανότητα η τουρκία να εκβιάσει και πάλι την ευρωπαϊκή ένωση εκτό από τι προσφυγικέ ροέ στα ελληνικά νησιά και την ιταλία. η ευρωπαϊκή ένωση κύριε μπορέλ δεν μπορεί να είναι ουραγός των εξελίξεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα ένα λεπτό. Η κυρία Εντσίρα από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπορέλ, είπατε ότι έγιναν κάποια βήματα και κάπου φάνηκε ένα πρώτο φως στο βάθος του τούνελ πείσαμε με την πτώση του Καντάφη ότι θα επέλθει δημοκρατία και ασφάλεια. Εγώ έχω επανειλημμένα επισκεφθεί και την περιοχή τα τελευταία χρόνια και υποστηρίζω τις δημοκρατικές δυνάμεις. Ε, βεβαίως η ελευθερία θα πρέπει να έρθει στη χώρα, αλλά τώρα τι έχει γίνει. Ε, Διώξαν ένα δικτάτορα και ήρθε το χάος. Δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπάρχει δημοκρατία και κενό εξουσίας είναι αυτό που επικρατεί εκεί. Η κατάσταση στη Λιβύη απαιτεί ε, κατάπαυση του πυρός που να τη σέβονται όλες οι πλευρές Μόνο έτσι θα επέλθει κάποια στιγμή μακροπρόθεσμα μια πολιτική λύση. Ε, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα ρόλο πολύ μεγαλύτερο για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών αξιών. Ε, η πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Λυπάμαι πάρα πολύ που σας κόβω το μικρόφωνο. Ο κύριος Ζορντάν ε, Μπαγντελά. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα σε πολλά μέρη του κόσμου. Δεν παίξαμε ρόλο ε, στη Συρία, δεν παίξαμε ρόλο στην επιδείνωση των σχέσεων Ιράν-ΗΠΑ ε, και δεν παίζουμε ρόλο και στη Λιβύη. Μόνο η Ρωσία και η Τουρκία βρίσκονται παρούσες εκεί. Το 2011 μερικοί δεν δίστασαν για ανθρωπιστικούς διθεν λόγους να πνίξουν στο αίμα την Λιβύη. Πώς λοιπόν να παίξουμε ρόλο. Ο κύριος Μπαρόσο, τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ζητούσε την εκδίωξη του Καντάφη, ε, καταστρέφοντας έτσι την χώρα που ήταν η πιο προοδευμένη σε όλη την Βόρεια Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η δική σας Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να μας κάνει πιο ισχυρούς, μας κάνει πιο αδύναμους πολλές φορές. Ε, τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμπίπτουν με τα συμφέροντα των λαών τη. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Αντιπρόεδρο, είπα το εκπρόσωπο κύριε Μπορέλ. Έχετε το λόγο για να κλείσετε. Άκουσα τα σχόλιά σας. Ε, πρέπει και εσείς να ζητήσετε από τον... Ε, μου λέτε πρέπει να ζητήσουμε την ακύρωση συμφωνίας Ερντοάν Σαράτς. Μπορώ να το ζητήσω. Και τι θα γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ήμασταν ποτέ ενωμένοι για τη Λιβύη. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς εδώ στην Ευρώπη ήμασταν διχασμένοι. Είχαμε αποκλίνουσες απόψεις. Και τώρα ενδεχομένως πληρώνουμε το τίμημα. Γιατί δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια ενιαία πολιτική προσέγγιση του ζητήματος. Είναι αλήθεια. Είναι κρίμα που η Τουρκία παίζει ρόλο. Αλλά ε, παίζει. Τι να κάνουμε. Και η Ρωσία το ίδιο. Σύμφωνα με τα τελευταία νέα, ο Χαφτάρ δεν υπογράφει την κατάπαυση του πυρός, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έπρεπε αν την υπογράψει να συμφωνήσει με την συμφωνία μεταξύ Σαράτζ και Τουρκίας. Όμως είπε ότι θα βρεθεί στο Βερολίνο την επόμενη Κυριακή. Ωραία. Η κακή είδηση είναι ότι δεν υπογράφει την ε, κατάπιση του πυρός. Η καλή είδηση είναι ότι παρόλα αυτά θα παραστεί στο Βερολίνο. και ίσως εκεί γίνει το πρώτο βήμα μιας πολιτικής συμφωνίας. Ίσως έχετε διαβάσει, έχετε παρακολουθήσει όλες μας τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις για τη Λιβύη στο, μετά το Σύμβουλο Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά και τις δικές μου. Ελπίζω, ας ελπίσουμε ότι στο Βερολίνο θα βρεθεί μια συμφωνία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, αλλά μετά θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας που θα απαιτήσει δύο πράγματα. Πρώτον, την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός. Δεύτερον, την, ε, τον έλεγχο του εμπάργου όπλων. Θα υποβάλω συγκεκριμένες προτάσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει πιο σημαντικό ρόλο σε αυτά τα δύο. Νομίζω ότι έχουμε την επαρκή αποφασιστικότητα να δράσουμε μαζί σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον και να ξεκινήσουμε μια καινούρια σελίδα στη Λιβύη. Αυτά μόνο μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Σχολιάσατε πολλές πτυχές του προβλήματος. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε όλους, σε όλες σας ερωτήσεις, αλλά μπορώ να συνοψίσω λέγοντας ότι αν προκύψει συμφωνία στο Βερολίνο, θα γίνει η κατάπιση του πυρός και τότε θα τεστάρουμε την πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να εμπλακεί περισσότερο στο, λιβικό, στο λιβανικό ζήτημα. Συγγνώμη, στο λιβικό ζήτημα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Ε, κλείνει έτσι αυτή η συζήτηση, αυτό το θέμα. Θα